Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας για να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία έχω να σας κάνω ε, δύο ανακοινώσεις. Η γραπτή δήλωση 47 σχετικά με τα ψάρια ως κοινό αγαθό συγκέντρωσε τις υπογραφές μεγαλύτερου αριθμού βουλευτών από την απλή πλειοψηφία του σώματος και κατόπιν αυτού θα διαβιβαστεί σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση, ενώ τα ονόματα των υπογραφόντων θα δημοσιευθούν στα συνοπτικά πρακτικά. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μίλανα εκ των συντακτών της γραπτής δήλωσης. Κύριε Μίλανα, έχετε το λόγο παρακαλώ. Grazie signor Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Αρσένη, την πεδρά Νέβες και Ρωμέβα και τους βοηθούς τους που συνεργάστηκαν ουσιαστικά για να πετύχει όλη αυτή η πρωτοβουλία. Τα Ψάρια είναι ένα κοινό αγαθό που δίνουν τεράστιο ποσοστό πρωτεϊνών σε ένα σωρό κόσμο και εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από την αλία. Πρόκειται για ένα κοινό δημόσιο αγαθό. Η έγκριση αυτής της δήλωσης υποδεικνύει στην Κομισιόν μία πορεία πολύ συγκεκριμένη για υπεύθυνη συμπεριφορά και των αλλιέων αλλά και των καταναλωτών. Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της αλλίας από σήμερα υποστηρίζει ακόμη περισσότερες δράσεις για την προστασία των αλλιευτικών πόρων και των εσωτερικών πολιτικών. Προτείνονται στρατηγικές για τη θάλασσα ως τον κατάλληλο χώρο για την αύξηση των αναπαραγωγικών της δυνατοτήτων και ως προς την αλληλευτική δραστηριότητα αλλά και μέσα από τις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και την προστασία της κοινωνικής οικονομικής συνοχής των αλλιέων και των οικονομιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιλάνα. Θέλω να σας ε, ενημερώσω ότι και η γραπτή δήλωση υπαριθμών 52 σχετικά με τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Down συγκέντρωσε τις υπογραφές μεγαλύτερου αριθμού βουλευτών από την απλή πλειοψηφία